Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω σε αυτή τη συνέντευξη τύπου με θέματα νέα ειδικά μέτρα για την Ελλάδα για τη διευκόλυνση της χρήσης και απορρόφησης ενωσιακών πόρων. Χαιρετίζω εδώ την παρουσία της κυρίας Μιχαήλοβα για την Περιφερειακή Επιτροπή και την κυρία Επίτροπο Κρέτσου που παρίσταται και αυτοί για να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις σας και για την παρουσίαση των νέων μέτρων. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για την προσέλευσή σας, για το ενδιαφέρον της Επιτροπής Περίφ. Σήμερα η Επιτροπή Περίφ είχε έκτακτη συνεδρίαση. Εκτός δηλαδή των τακτικών μας συνεδριάσεων η πρώτη θα είναι τη 17η Σεπτεμβρίου. Από όλοι οι συντονιστές λοιπόν της Περιφερειακής Επιτροπής ε, συμφώνησαν να οργανωθεί η αυτή έκτακτη συνεδρίαση διότι λόγω των προτάσεων της Κομισιόν για την ε, διόρθωση μετατροπή του κανονισμού για την Ελλάδα και επομένως όλοι μαζί τα μέλη της Επιτροπής, το Προεδρείο, οι συντονιστές καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να γίνει μια συζήτηση ώστε να διασφαλιστεί ότι θα καταλαβαίνουμε καλά τι λέει η πρόταση, να συναντήσουμε την Επίτροπο, να ακούσουμε όλες τις εξηγήσει που έχει να μας δώσει για τους λόγους που γίνεται αυτή η τροποποίηση του κανονισμού και τα μέτρα που προτίθεται να λάβει στο μέλλον για να ελεγχθεί η κατάσταση. Ήταν πολύ καρποφόρα συνάντηση λοιπόν. Σχεδόν όλα τα μέλη που προσήλθαν έλαβαν και το λόγο πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση διότι όλα τα μέλη συμφώνησαν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και η πολιτική συνοχής για να στηριχθεί η οικονομία της Ελλάδας και η διαβίωση των πολιτών της. Όλοι οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο ανέφεραν τη σημασία της απόφασης αυτής, όλοι ανέφεραν τη σημασία του ελέγχου της εφαρμογής αυτής της απόφασης στο μέλλον διότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αυτά τα χρήματα θα πάνε άμεσα, θα διατεθούν άμεσα σε σημαντικά προγράμματα και σχέδια, θα ελέγχεται η εφαρμογή τους και θα υποβάλλονται τα συμπεράσματα των ελέγχων αυτών και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο. Αποφασίσαμε λοιπόν τελικά ότι η καλύτερη λύση για μας στο Κοινοβούλιο είναι να ακολουθήσουμε μια απλή διαδικασία που υπάρχει ήδη από τον κανονισμό του Κοινοβουλίου το άρθρο 50 του κανονισμού του Κοινοβουλίου και συμφωνήσαμε μόνο ένα μέλος απήχε όλοι οι υπόλοιποι υποστήριξαν το, τη διαδικασία αυτή χειρισμού των προτάσεων της Κομισιόν. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη, άκουσα πολλές ιδέες για τον ρόλο της Επιτροπ... Περιφερειακής Επιτροπής για καλύτερο συντονισμό με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών και της Επιτροπής μας και είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να βρούμε έναν βέλτιστο τρόπο ελέγχου της διαδικασίας αυτής, παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της και για να δούμε πώς μπορούμε να σταματήσουμε την εφαρμογή όχι βελτίστων πρακτικών σε μερικές χώρες τουλάχιστον γιατί εμείς στην περιφερειακή καταλαβαίνουμε ότι αφορά με την Ελλάδα η απόφαση αλλά επίσης θα έχει επιπτώσει στην περιφερειακή πολιτική γενικότερα και την εφαρμογή της σε όλες τις χώρες μέλη. Πολύ χρήσιμη λοιπόν η συνάντηση, πολύ καλή η συζήτηση και καλή συνεργασία με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ παρόντε. Χαίρομαι που είμαι εδώ με την Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερική Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου και την, δηλαδή την κυρία Ίσκρα Μιχαηλόβα. Ευχαριστώ πολύ για την προσωπική σας εμπλοκή, για την επιτυχία που συνοδεύει τη σημερινή μας συνεδρίαση. Όπως είπε η κυρία Πρόεδρος πιο πριν, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να βοηθηθεί να συνδραμεί η Ελλάδα να μπορέσει να προχωρήσει με τα διαθωτικά και τα επενδυτικά προγράμματα και κονδύλια και με την παρουσίαση αυτών των μέτρων μέσα από τις δράσεις τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και την Δημιουργία Απασχόλησης στην Ελλάδα στις 15 Ιουλίου, κατά το 2014 στο 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 35 δις θα επενδύσει στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων 20 δις από τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία για την ανάπτυξη. Και φυσικά πρόκειται για χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με αυτά τα κονδύλια. Είναι σημαντική συνεισφορά για την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας, της ε, περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής σε αυτές τις δύσκολες ε, χρονικές στιγμές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να υπάρξει η διάνοιξη μιας θετικής προοπτικής για το μέλλον της Ελλάδας η πρότασή μας ε, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα όσον αφορά τα θέματα της πολιτικής συνοχής για την Ελλάδα. Αυτά τα μέτρα τώρα είναι στα χέρια πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να προχωρήσουν και να ευδοκιμήσουν των νομοθετών δηλαδή. Και όπως επεξήγησα τους Ευρωβουλευτές δεν μπορώ να τονίσω επαρκώς την σπουδαιότητα του να εγκριθούν αυτά τα έκτακτα μέτρα το δυνατόν νωρίτερα και είμαι το δυνατόν νωρίτερο και είμαι πραγματικά ε, ευγνώμων για την ε, σχεδόν ομοφωνία που επετεύχθη σήμερα στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου διότι αυτά τα κονδύλια πρέπει τώρα να απελευθερωθούν ώστε να μπορέσουν νέα κονδύλια να ρεύσουν και να υποστηρίξουν τις ε, επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της Ελλάδας. Λέγοντας αυτά, έκτακτα μέτρα είναι σημαντικά και για το, ε, την περίοδο 2007-2013 καθώς επίσης και για την περίοδο 2014-2020 για τις δράσεις των κονδυλίων αυτών. Από το 2014 στο 2020 προτείνουμε να αυξηθεί το ποσοστό της αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα συνοχής ε, κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό το μέτρο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο και θα δώσει τη δυνατότητα πρόσθετα κονδύλια να διατεθούν επί δύο έτη. 500 εκατομμύρια το 2015 και 500 εκατομμύρια το 2016 ε, για την προλίανση των δραστηριοτήτων. Για την περίοδο 2007-2013 ε, προτείνουμε το τελευταίο 5% των πληρωμών που ουσιαστικά θα παρακρατούν το μέχρι την ολοκλήρωση και το κλείσιμο λογαριασμό το 2017 άμεσα να διατεθούν στις ελληνικές αρχές, στην ελληνική κυβέρνηση. Επίσης ε, προτείνουμε να αρθεί η ανάγκη, η ρήτρα εθνικής χρηματοδότησης, ε, ώστε το ποσοστό 100% χρηματοδότησης να μπορεί να ισχύει για την περίοδο του 2007-2013. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρόσθετα 500 εκατομμύρια θα διατεθούν άμεσα κιόλα μετά τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όταν επιτευχθεί. Αυτό επίσης θα ανακουφίσει την πίεση στον προϋπολογισμό προπολογισμό, τον ελληνικό προπολογισμό, κατά 2 εκατομμύρια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια τώρα σε σχέση με την προχρηματοδότηση είναι κάτι το οποίο στον εθνικό προπολογισμό θα αντανακλάται. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται εκ του σύνεγγυ με τι ελληνικέ αρχέ ώστε να επιτεθούν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα διαρθρωτικά και επενδυτικά κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο θέμα τη δαπάνη, τη διάθεση των κονδυλίων, αλλά τη διάθεσή του με συνετό και αποτελεσματικό τρόπο. Με στοχοθετημένα μέτρα ώστε να υπάρξει σε ανάκαμψη και ανάπτυξη όπως την έρευνα και ανάπτυξη ή την υποστήριξη για την ανάπτυξη <clears throat> και την ε, δυνατότητα να διανοιχτούν ε, στον διεθνή ανταγωνισμό οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι μια απόδειξη της αλληλεγγύης που πάντα καταδεικνύαμε, δείχναμε έναν της Ελλάδας με οικονομική και νομική υποστήριξη και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτή τη βοήθεια και στο μέλλον. Φυσικά ήμουν και έχω επισκεφθεί την Ελλάδα και θα ξαναπάω στην Ελλάδα και πάλι, ώστε να μπορέσουμε σε ανταλλαγή απόψεων με του εμπλεκόμενου να εκθέσουμε το τι γίνεται και μπορεί να γίνει με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τις ελληνικές αρχές για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σχόλια και ερωτήσει. Να λέτε και το όνομα και την ιδιότητά σας και Δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, υπάρχει κανένας οδικός χάρτης, κανένα πρόγραμμα για την αποφυγή των κακών πρακτικών όπως μπορεί να μειώνονται στην Ελλάδα. Δεύτερον, 35 δις θα επενδυθούν στην Ελλάδα τα 13 από τα διαρθρωτικά ταμεία μπορεί να επικαλύπτονται με προγράμματα όπως τον ορίζοντα 2020 ή μήπω όχι. Καταρχήν για την εφαρμογή αυτό είναι πάντα ευθύνη των χωρών μελών. Οι ελληνικές αρχές λοιπόν νομίζω ότι γνωρίζουν ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε την Ελλάδα, αλλά φυσικά έχουν και αυτοί υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα να δημιουργήσουν αυτά τα διοικητικά σώματα που πρέπει να ταυτίζουν τα υψηλής ποιότητας προγράμματα και σχέδια και πάντα όσα επαναλαμβάνω τέτοια πράγματα είναι ευθύνη των χωρών μελών. οι κακές πρακτικές υπάρχουν παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και οι διοικητικέ δυνατότητες είναι πολύ σημαντικές. Πιο σημαντικές και από τα χρήματα νομίζω. Γιατί πολλές χώρες υπάρχουν που περιμένουν να πάρουν χρήματα από τις Βρυξέλλες. Οι Βρυξέλλες περιμένουν να τους δώσουν χρήματα αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα διοικητικά να τα απορροφήσουν αυτά λοιπόν πάνε χέρι με χέρι, τεχνική βοήθεια, χορήγηση χρημάτων και υποβοήθηση τη λειτουργία του Υπουργείου Οικονομικών για ορισμένα θέματα όπου υπάρχουν αδυναμίες στις δημόσιες προμήθειες και άλλα και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή του είδους η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Κομισιόν. Όσο για τα 35 δις, τα 20 προέρχονται από τα διαρθρωτικά και παιδιτικά ταμεία και 15 άμεσα για τους γεωργούς. Αυτά όλα είχαν προβλεφθεί για την Ελλάδα στο πρόγραμμα μέχρι το 2020. Τώρα όμως λέμε να τα χορηγήσουμε νωρίτερα, front loading 15 με 20 με 15 με 16 ώστε να μπορέσει να λυθεί αυτό το πρόβλημα εφόσον μάλλον λυθεί αυτό το πρόβλημα της ε, απορροφητικότητας. Βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από αυτά που θα έχει εγκρίνει και εφαρμόσει η Ελλάδα στη συμφωνία. Ελπίζω λοιπόν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις τους τα επόμενα δύο-τρία χρόνια μαζί με τη δική μας πρόταση θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο στην ελληνική οικονομία και για τον ελληνικό λαό και για την περίοδο μέχρι το 30 γνωρίζετε ότι ο κίνδυνος αν δεν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα είναι πολύ ψηλός διότι όταν εγώ ανέλαβα τα καθήκοντά μου η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που είχαν 90% απορρόφηση και τώρα έχει μειωθεί κατά πάρα πολύ. Ο κίνδυνος όμως ήταν ότι δεν είχαν ε, ότι δεν υπάρχει ρευστότητα και γι' αυτό για να οικοδομηθεί ένας αυτοκινητόδρομος ας πούμε αν δεν εγκριθούν αυτά τα μέτρα σήμερα δεν θα μπορεί η Ελλάδα να προσφέρει να συνεισφέρει το 5% για τον αυτοκινητόδρομο και θα υποχρεωθεί να επιστρέψει όλα τα χρήματα για μη συμπλήρωση του προγράμματος. Είναι λοιπόν μια ιστορική σημασία ε, χειρονομία αλληλεγγύης που κάναμε για την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω δύο λόγια εμείς στην Επιτροπή Περιφερικής Ανάπτυξης είμαστε στεναροί υποστηρικτές της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει πρόταση για οποιασδήποτε αλλαγές στα πολιετή δημοσιονομικά πλαίσια. Εργαστήκαμε με την ενισχύ νομοθεσία και κανονισμούς και διατάξεις, με, το ενισχύ, με τις ενισχύ ευκαιρίες για την Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό δεχθήκαμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν τροποποιεί οποιασδήποτε άλλες δυνατότητες για τις άλλες χώρες δημοσιονομικά. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Εργαζόμαστε με τις ευκαιρίες που παρέχονται στην Ελλάδα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να προωθήσουμε, να προαγάγουμε κάπως, να υποστηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τις πληρωμές στο τελευταίο έτος της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή του 2007-2013, για να κλείσουν. Αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο υποστηρίζουμε αυτή την πρόταση και δεύτερον, όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής αναφέρουν αυτό το οποίο λέγεται στο τέλος αυτής της πρότασης, ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει, υποτίθεται θα ακολουθήσει και θα συμμορφωθεί με όλους τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Και αν δεν ε, γίνουν ε, όλα αυτά και δεν χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες να χρησιμοποιηθούν αυτά τα επιπλέον κονδύλια, θα επιστραφούν. Είναι υποχρέωση να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά είναι δύο σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα, μεγάλη σημασία σε αυτή την πρόταση. Δίνουμε ευκαιρία στη χώρα, στην Ελλάδα, να ανακάμψει. Ταυτόχρονα όμως αυτό που κάνουμε είναι ακολουθούμε και συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες που είναι ίσοι και ίδιοι για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μεγάλη σπουδαιότητα. Σε ευχαριστώ. Άλλε ερωτήσεις παρακαλώ. Um, Υπάρχει κανένα πρόγραμμα για τη λήψη της τελικής απόφασης για την έγκριση των πολιετών προοπτικών από το κοινοβούλιο ας πούμε. Όχι, για αυτά τα μέτρα, όχι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Α, ναι, με συγχωρείτε. Είπα ότι δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Άλλο τα μέτρα. Έχουμε κάποιον οδικό χάρτη, πολύ σύντομο. Δηλαδή συζητήσαμε πώς θα γινόταν αυτό με το πιο εύκολο και γρήγορο δυνατό τρόπο η ομάδα εργασίας συναντήθηκε και με εκπροσώπους του Συμβουλίου, θα ξανασυναντηθούν με αύριο και θα μάθουμε τι φρονεί το Συμβούλιο, ποια είναι η απόφαση του Συμβουλίου και μετά στην Περιφερειακή Επιτροπή θα κάνουμε την τακτική μας συνεδρίαση στις 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού θα, αν αυτή η πρόταση θα το υποβάλω στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, δηλαδή στην Ολομέλεια. Αυτό είναι το πρόγραμμα, πολύ σύντομο. Γιατί αποφασίσαμε αυτό να ακολουθήσουμε, τη γρήγορη διαδικασία. Συζητήσαμε επίσης στην Περιφερειακή Επιτροπή να συνεργαστούμε στενότερα με τα κράτη-μέλη είπαμε να καλέσουμε πολλούς υπουργούς από διάφορες χώρες, ιδιαίτερα από τις χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα. Θα καλέσουμε λοιπόν και τον Έλληνα Υπουργό που θα είναι υπεύθυνο για την συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη και θα είναι μια πραγματική συζήτηση για το πώς θα γίνει η εφαρμογή γιατί η Κομισιόν έκανε την πρόταση, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την πρόταση της Κομισιόν, μάλλον θα, το ίδιο θα κάνει και το Συμβούλιο και τώρα το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μένει να δούμε τι θα κάνει. Έτσι θα παρακολουθούμε την εφαρμογή των μέτρων. Τελευταία ερώτηση, ορίστε. Μαρία Ρόνια από την Athens News Agency είπατε ότι προτείνατε την προχρηματοδότηση, υποκαταβολές δηλαδή χρηματοδότησης για το ποσό αυτό το 2015 και 2016 όπως αναφέρατε. Υποθέτω ε, ότι έχετε ήδη ίσως ταυτοποιήσει κάποια συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς και ποια είναι αυτά και ποιοι είναι αυτοί οι τομείς. Είπατε ότι κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην Ελλάδα είπατε ότι θα επισκεφθείτε το φθινόπωρο την Ελλάδα. Ποιες περιοχές, ποιες περιφέρειες θα επισκεφθείτε στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η κυρία Μιχαηλόβα πιο πριν, είναι ουδέτερο ε, χωρί δημοσιονομικέ άλλε επιπτώσεις ή στρεβλώσεις αυτό ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις προχρηματοδοτήσει, Θέλουμε απλώ να καταβάλουμε κονδύλια ταχύτερα, αλλά δεν πρόκειται για επιπρόσθετα ξεχωριστά κονδύλια. Σύμφωνα με τον, χρονο, τον οδικό χάρτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και όσα έχουν προβλεφθεί ελπίζουμε ότι τον Οκτώβριο ή ήδη δηλαδή τις πρώτες ε, καταβολές ε, ε, ρευστότητας με αυτά τα κονδύλια, την τόνωση ρευστότητα στην Ελλάδα με αυτά τα μέτρα. Και όπως είπα για το 2014-2015 θα είναι ένα δισεκατομμύριο και στη συνέχεια άλλο ένα δισεκατομμύριο. Δύο δισεκατομμύρια δηλαδή συνολικά που θα ανακουφίσουν τον ελληνικό προϋπολογισμό. Αυτά είναι ήδη τα πρώτα βήματα και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε αποτελεσματικοί. Ότι δηλαδή εμένουμε και επιμένουμε στο κατεπήγον της έγκρισης λοιπόν και την ταχύτητα έγκρισης αυτών των μέτρων για να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Αν Οκτώβριο είναι ήδη με καθυστέρηση η ημερομηνία. Αν θέλουμε να έχουμε επιπτώσει στην ε, πραγματική οικονομία, πρέπει να δράσουμε αμέσω. Ξέρουμε ότι η περίοδο 2007-2013 λύγει η περίοδο αυτή το Δεκέμβριο 2015. Λοιπόν, αν ίσχυαν οι κανονικέ διαδικασίε, αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν να διατεθούν στην Ελλάδα. Δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στην πραγματική ελληνική οικονομία. Εγώ επισκέφτηκα την Ελλάδα. Αληθεύει αυτό. Το γνωρίζετε καλά και το είπα και πριν από πέντε ημέρες είχα επαφές με υπουργούς. Επισκέφθηκα τέσσερις περιφέρειες, τέσσερις περιοχές. Συνάντησα όλους τους ε, διοικητές, ε, τους περιφερειάρχες και νομίζω ότι κατανοούν καλύτερα πώς λειτουργούν και αλλάζουν το πρόσωπο, το χαρακτήρα της Ελλάδας στα διαθωτικά ταμεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, μετά δηλαδή την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες επιπτώσεις είχαν αυτά τα κονδύλια. Κάνω λόγο για τα επενδυτικά και τα διαθωτικά κονδύλια. Μέσα σε αυτά τα 34 χρόνια 73 δις εισήχθησαν ως ένεση στην ελληνική οικονομία και επιπρόσθετα μέτρα τόνωσης και ανακούφισης. Αν δούμε το πρόσωπο, την εικόνα της Ελλάδας πριν από τη δεκαετία του 80 μπορεί κανείς να αντιληφθεί άμεσα πόσες μεγάλες αλλαγές έγιναν και επισκέφθηκα πολλά τέτοια προγράμματα και σχέδια και η γέφυρα που Ρίου Αντιρίου που συνδέει τη στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο και όσα έγιναν και σε σχέση με το μετρό και άλλες δραστηριότητε. ήταν μεγάλες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δισεκατομμύρια για την Αθήνα και για το μετρό τον υπόγειο της, ε, των Αθηνών. Κανόνα λόγο λοιπόν για τι αλλαγέ αυτέ που τα ευρωπαϊκά κονδύλια συνεισέφεραν να επιτευχθούν με μεγάλη χαρά είδα ότι στι περιφέρειε ιδιαίτερα κατανοούν πολύ καλά τον ρόλο των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων οι πολίτε, Το τι έγινε δηλαδή κατά τα τελευταία 35 χρόνια. Από ό,τι γνωρίζω εγώ με τον Υπουργό ε, Σταθάκη για την Οικονομία έχω, είχα επαφέ και είναι σαφέ ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει σε σχέση με τις, ε, ε, την επίσπευση των εκλογών να δούμε πώς θα μπορέσει να ε, λειτουργήσει. Και με την νέα υπηρεσιακή κυβέρνηση έχουμε συνεργασία. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστούν αυτά τα μέτρα άσχετα από το θέμα των εκλογών. Είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων, του ελληνικού λαού να γίνει αυτό και να προχωρήσουν. Θα υπήρχε μια μεγάλη διάσκεψη για την έρευνα και διάσκεψη και τις την εξειδίκευση. Θα είμαστε σε επαφή από πλευρά γραφείου μου με την Ελλάδα και εσάς και θα σας γνωστοποιήσουμε Πότε θα γίνει αυτό. Η ιδέα μας είναι να έχουμε αυθεντικούς εταίρους ώστε να γίνει συζήτηση και διαβούλευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αλλά θα πρέπει ταχύτατα να γίνουν αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αναβαθμισμένα υψηλή ποιότητα τέτοια προγράμματα και σχέδια που θα προαγάγουν τις θέσεις απασχόλησης και την ε, ε, πρόοδο και την ανάκαμψη της Ελλάδας. Για τους νέους ιδιαίτερα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι πολύ γνωστό αυτό και φυσικά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε επίσης και για τα θέματα μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά. Είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο προσβλέπουμε να συζητήσουμε με τις αρχές, με την κυβέρνηση και τη διοίκηση στην Ελλάδα. Εξετάζουμε και βλέπουμε πώς ε, τα δικά μας κονδύλια θα μπορούσαν να συνεισφέρουν επίσης να ανακουφιστεί η κατάσταση σε σχέση με την μετανάστευση. Η Ιταλία για παράδειγμα παράδειγμα, χρησιμοποίησε πολλά κονδύλια από το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα θέματα μεταναστών και στην Απουλία, Πούλια και σε άλλες περιοχές. Και θα πρέπει εδώ να δούμε την δυνατότητα για την Ελλάδα τέτοιου είδους κονδύλια να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για δράσεις και σχέδια. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και την Ελλάδα λοιπόν με ταχύτατες δράσεις σε αυτή την κρίση, ανθρωπιστική κρίση που πλήττει, που μαστίζει την Ελλάδα με τα θέματα της μετανάστευσης μετανάστευσης δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελείωσε ο χρόνος μας.